was closed. Okay, very good. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ήρθε η προσκεκλημένη μας. Βρήκε και την κρυφή αίθουσα. Την ανακάλυψε, λοιπόν. Ρίξουμε μια ματιά στην ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να αλλάξει κάτι δεν μου έχουν πει τίποτα οπότε μπορούμε να περάσουμε το σημείο 1 σημείο 2 ανακοινώσει του Προέδρου έχω να πω το εξής ε, συναντήθηκαν οι συντονιστές αυτή την εβδομάδα για να αποφασίσουν το εάν θα μείνει η επίσκεψη στην Αθήνα όπως έχει ή μήπως θα αναβληθεί γιατί μάθαμε ακριβώς τη μέρα της επίσκεψής μας που θα συναντηθούμε 9 η ώρα με τους εκπροσώπους των συνδικάτων. Σε 11 η ώρα ξεκινάει 24ωρη γενική απεργία. Έχει αποφασιστεί ήδη από τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα που εκπροσωπούν συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους. Οπότε, είπαμε, καλύτερα να γίνει μια αναβολή, το συζητήσαμε με τους συντονιστές και κατά πλειοψηφία λάβαμε, δημοκρατικά ψηφίσαμε ε, και λάβαμε την απόφαση να αναβάλουμε το ταξίδι κατά ένα μήνα. Θα γίνει 22 και 23 Μαρτίου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό βεβαίως και έχουμε καλές πιθανότητες να βρούμε υψηλόβαθμους συνομιλητές οπότε υποθέτω πως ε, η επίσκεψη θα είναι επικοδομητική αλλά ως πρόεδρος δεν θα ήθελα να βρεθούμε στη μέση μιας γενικής απεργίας να μην υπάρχουν και αντιπαραθέσεις και να αποτελέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικείμενο μιας εσωτερικής ελληνικής ε, αντιπαράθεσης. Αυτά λοιπόν για αυτό το θέμα. Τώρα καλωσορίζω την κυρία Ελένα Φλόρες Γουάλ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δήλωσε να ε, διατεθειμένη να κάνει μια εισαγωγή στο θέμα αυτό για να δούμε πώς θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα την αηφορία της οικονομίας και όλα αυτά με βάση το ότι έχουμε μια φιλόδοξη και απαιτητική στρατηγική για την Ευρώπη 2020. Ξέρετε πως πρέπει να καταφέρουμε τουλάχιστον να βρεθούμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης. Εάν δεν τα καταφέρουμε, τότε δεν θα είναι μόνο θέμα εκπλήρωσης στρατηγικής 2020, αλλά θα έχουμε και δυσκολίες με το δημόσιο χρέος και τη μείωσή του και έτσι η κρίση του ευρώ δεν θα έχει λυθεί αλλά θα μας συνοδεύσει για χρόνια και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να είναι στο προς το συμφέρον κανενός κράτους μέλους, ανεξαρτήτως του εάν έχει ταλαιπωρηθεί ο προϋπολογισμός του ή όχι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και χαίρομαι για το ότι παρά το ότι είναι πέμπτη απόγευμα είναι αρκετοί συνάδελφοι εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν ας ακούσουμε την κυρία Φλόρες. Ε, αν μπορείτε να μας δώσετε μια γενική εικόνα σε 10-12 λεπτά και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Uh, apologize. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Κοιτάξτε, και το γραφείο μας είναι λίγο μακριά από εδώ και είχε κλείσει και η κυρία είσοδος, οπότε χαθήκαμε στο κτίριο που προσπαθούσαμε... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ επίκαιρη συζήτηση αυτή και πρέπει να σας πω ότι από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό που σκοπεύω να κάνω είναι, όπως είπε ο πρόεδρο, να σας κάνω μια σύντομη εισαγωγή, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να ακούσουμε τι έχετε να πείτε εσείς και θα ήθελα να ακούσω και εγώ τι θέλουν να πούνε οι βουλευτές, που εντοπίζετε τις προτεραιότητές σας, που εντοπίζετε αδυναμίες. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για να προχωρήσει η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και όλες οι πρωτοβουλίες που έχουν τεθεί θα τεθούν επιτάπητος. Επομένως, με βάση αυτό που σας προείπα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και ελπίζω να έχουμε χρόνο ώστε και να σα ακούσω και να κάνω και κάποια σχόλια. Όπω είπε ο πρόεδρο, Έχουμε μια πολύ φιλόδοξη στρατηγική καταθέσει, τη λεγόμενη στρατηγική για την Ευρώπη 2020. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι τόσο το όνομα, ο τίτλος, αλλά το περιεχόμενο η ουσία, οι πολιτικέ δηλαδή που πρέπει να εφαρμοστούν. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να εστιάσουμε στι πολιτικέ. Και το λέω αυτό γιατί ενίοτε έχω την εντύπωση και αληθεύει κιόλα νομίζω ότι υπάρχουν τόσε πολλέ πρωτοβουλίε με τόσα πολλά ονόματα κτλ. που τα χάνουμε λίγο. Ο κόσμο ε, ε, συγχαίει ορισμένα πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μα τι είναι σημαντικό. Και το περιεχόμενο των πρωτοβουλειών πρέπει να είναι συμπληρωματικό και συνεπές και έτσι μπορούμε να δούμε όλες αυτές τις προτάσεις. Πού βρισκόμαστε λοιπόν και προς τα πού οδεύουμε. Είναι προφανές ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει. Η πραγματική οικονομία βέβαια αρχίζει να ανακάμπτει, ε, να βελτιώνεται, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ μικρή η πρόοδος και υπάρχει, υπάρχουν πολύ κίνδυνοι ακόμη. Έχουμε κάποια θετικά σημάδια βέβαια, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Γνωρίζουμε ότι εάν δεν λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο μεταρρυθμίσεων και αν δεν εστιάσουμε στις πολιτικές μας ε, η ανάκαμψη θα είναι άτολμη και δεν θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας. Ε, γι' αυτό λοιπόν και έχοντας υπόψη τις ανησυχίες και τα γεγονότα αυτά, γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η στρατηγική ανάπτυξη. Τρεις πτυχές νομίζω αξίζει να υπογραμμίσω εδώ. πρώτα απ' όλα παγίωση δημοσίων οικονομικών και εξυγίανσή τους ε, δεν είναι κάτι που μας αρέσει και το λέμε απλά έτσι, απλά ε, είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα κράτη-μέλη για δύο λόγους. Πρώτο γιατί η κρίση έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη μείωση των ε, εσόδων, όπως είναι φυσιολογικό σε αυτή την κυκλική ε, φάση, αλλά αυξάνουν οι κυβερνήσει ταυτόχρονα τι δαπάνε για να αντιμετωπίσουν την κρίση και αυτό οδήγησε και πολλέ φορέ σε αύξηση πολύ μεγάλη του ελλείμματο και συσσόρευση χρέου. Εδώ λοιπόν για πολύ καλού ε, λόγου, για βάσιμους λόγου, καλού και κακού. έχουμε αυτή την κατάσταση, δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση αυτή το γνωρίζουμε με τις αναλύσεις που έχουμε κάνει και λόγω των δυσκολιών βέβαια που αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες για να βρουν κάποιον ο οποίος θα χρηματοδοτήσει το χρέος. Γι' αυτό και νομίζουμε ότι η δημοσιονομική εξυγένση είναι ένα από του τρει άξονε. Δεύτερον, είναι πιο βαθιά μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα. Έχουν γίνει πολλά πράγματα, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει την πορεία μας. Και τρίτον, Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε τι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει, Μεταξύ αυτών που πρέπει να γίνουν ε, για τι οικονομίε και είναι πολλά αυτά, πρέπει πια να επιλέξουμε τι πρέπει να γίνει πρώτο. Πρέπει να ιεραρχήσουμε τι προτεραιότητε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν και τα υπόλοιπα, αλλά υπάρχουν κάποια ε, πράγματα που είναι σημαντικότερο να γίνουν στην αρχή γιατί μπορούν ε, να προωθήσουν την ανάπτυξη και βέβαια μετά θα συνδυαστούν και με τις υπόλοιπες πτυχές που θα ακολουθήσουν. Με βάση αυτό το υπόβαθρο νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιπαρατάξει μια συνολική απάντηση στις τρεις αυτές προκλήσεις. Έχουμε τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, το πακέτο Οικονομική Διακυβέρνηση και Συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτά είναι τα τρία που θέλω να αναφέρω. Ξεκινήσαμε λοιπόν στις 12 Ιανουαρίου με την δημοσίευση της ετήσιας έρευνας για την ανάπτυξη που ουσιαστικά είναι συνέχεια της προσέγγισής μας στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και πρόθεσή μας με αυτή την έρευνα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που σας προείπα, δηλαδή να σταχυολογήσουμε τις βασικές προτεραιότητές μας, ε, γιατί θα υπάρξει και του χρόνου ετήσια έκθεση ανάπτυξης και θα δούμε τότε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες που θα επιλέξουμε. Δέκα δράσεις προτεραιότητας έχουμε που δεν θα τις ε, αναφέρω γιατί τις ε, περιλαμβάνει η έκθεση αλλά ομαδοποιούνται γύρω από τρεις βασικούς τομείς δημοσιονομική εξυγίανση, μακροοικονομική σταθερότητα μεταρρυθμίσει αγοράς εργασίας για μεγαλύτερη απασχόληση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Οι δέκα λοιπόν προτεραιότητες ομαδοποιούνται γύρω από αυτές τις τρεις βασικές πολιτικές, τους τρεις τομείς πολιτικής προανέφερα. Αυτή η αιτήσια λοιπόν έρευνα για την ανάπτυξη θα έλεγα ότι αποτελεί ε, το εφαλτήριο για το τι περιμένουμε να μας προτείνουν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ανταπόκρισή τους στις πολιτικές προτείνουμε. Τι θα πει αυτό αυτό που περιμένουμε από τα κράτη-μέλη, μάλλον το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περιμένουμε να δώσει κάποιες κατευθύνσεις για τις προτεραιότητες πολιτικής και βέβαια αναμένουμε οι προτεραιότητες αυτές, οι κατευθυντήριες γραμμές να συμβαδίζουν, να συνάδουν με αυτά τα οποία εμείς παρουσιάζουμε στην ετήσια έρευνα. Ίσως να υπάρχουν διαφορετικές επιλογές, θα το δούμε αυτό αλλά περιμένουμε από τα κράτη-μέλη συνεχεία στο πλαίσιο των στρατηγικών τους, δηλαδή προϋπολογισμοσχέδια αρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κυρίως, να ε, προχωρήσουν, να δώσουν μια συνέχεια στις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να δούμε συγκεκριμένα τι θα κάνουν το 2011 οι χώρες και επίσης να δούμε τι θα περιλαμβάνει και ο προπολογισμό του 2012. Αυτό περιμένουμε από τα κράτη-μέλη. Δεν θα εστιάσω σήμερα στη δημοσιονομική πλευρά γιατί νομίζω ότι ε, η φύση της συζήτησης είναι περισσότερο για τα άλλα ζητήματα, διαρθρωτικές πολιτικές για την ανάπτυξη θα έλεγα κυρίω. Και μπορώ να πω ότι έχει χαρτογραφήσει μια φιλόδοξη ατζέντα η Κομισιόν στο πλαίσιο τη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Θα δούμε κατά πόσο θα υπάρξει αποτελεσματική κινητοποίηση και επανεστίαση όλων των εργαλείων και μέσων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και βέβαια τα οριζόντια ε, εργαλεία είναι ο βασικό κινητήριο μοχλό, όπω είναι η αγορά επανεστίαση του κοινοτικού προϋπολογισμού και προβλεπτική χρήση εξωτερικών πολιτικών. Για το υπόλοιπο του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου ε, θα ήθελα να αναφέρω κάποιες από τις σημαντικές πολιτικές που νομίζω ότι πρέπει να ενεργοποιήσουν. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε απαραίτητη προσπάθεια για να αξιοποιήσουμε το πλήρε δυναμικό τη νέα αγορά. Είναι μια από τι βασικέ προτεραιότητε, εμβάθυνση τη νέα αγορά που θα έχει πολύ σημαντική θετική επίπτωση. Νομίζω ότι καλό είναι να επικεντρωθούμε σε λίγε δράσει που θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πλήρη υλοποίηση τη οδηγία για τι υπηρεσίε, την ολοκλήρωση του πλαισίου για την πνευματική ιδιοκτησία να έχουμε κάποια πρότυπα διαλειτουργικά ιδίω στους ε, τεχνολογίες πληροφοριών ε, και επικοινωνιών και κίνητρα για εμπόριο και επενδύσεις. Νομίζω ότι στο σκέλος ενή αγορά πρέπει να έχουμε εκεί πρόοδο πολύ γρήγορα. Στα περισσότερα από αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη διατυπώσει τις προτάσεις της και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα είναι ε, πλέον να πιέσουμε ώστε να εφαρμοστούν όλες αυτές οι προτάσεις. Σε ό,τι αφορά το πρώτο που ανέφερα, την οδηγία δηλαδή για τις υπηρεσίες, ο στόχος ήταν να έχει υλοποιηθεί έως τα τέλη του 2009 από τα κράτη-μέλη αυτή η οδηγία και στόχος μας είναι οι φορείς παροχής υπηρεσιών να μπορούν να εγκατασταθούν από τη μία χώρα στην άλλη, να μπορούν να παρέχουν διασυνοριακώς τις υπηρεσίες τους. Θα φροντίσουμε λοιπόν να εφαρμοστεί ορθά η οδηγία και να βελτιώσει τις υπηρεσίες και το εμπόριο. Θα επαγρυπνούμε επίσης για να μην αναδυθούν νέα ρυθμιστικά εμπόδια που θα αντικαταστήσουν αυτά τα οποία ήρε η οδηγία. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν μέτρα στον τομέα των πολιτικών που θα εξασφαλίσουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Εδώ νομίζουμε ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καινοτομία, στην οικονομία της γνώσης. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό βέβαια, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Κάναμε κάποιες εκτιμήσεις ε, και όχι μόνο εμείς, η Κομισιόν, αλλά και από κάποιες εξωτερικές μελέτες και από ε, πανεπιστήμια. Έχουμε κάποιες μελέτες λοιπόν για το όφελος ε, που συνεπάγεται η επένδυση στην καινοτομία και την οικονομία της γνώσης και μπορώ να σας αναφέρω ένα στόχος επενδύσεων του 3% του ΑΕΠΑ, έρευνα τεχνολογία μέχρι το 2020, θα δημιουργήσει 3,5 και παραπάνω εκατομμύρια θέσεις εργασίας. 800 δις ευρώ μέχρι το 2025. Ε, κάποιες αδρές εκτιμήσεις σας ε, κάνω τώρα. Υπάρχουν και άλλες μελέτες. Πάντως ε, σε αυτά τα νούμερα περίπου κινούμεθα. Είναι σημαντικό λοιπόν. Και για το σκοπό αυτό η πρωτοβουλία Ένωση της Καινοτομίας που θα τη βρείτε και στρατηγική 2020 εστιάζει σε διάφορες πτυχές καινοτομία, ε, οικονομία της γνώσης. Πρώτα απ' όλα αύξηση των επενδύσεων στα επίπεδα άλλων ηγετικών οικονομιών, μεγαλύτερα κίνητρα για τους επιχειρηματίες για να δώσουν ιδέες στις αγορές και άλλα πράγματα όπως καλύτερη πρόσβαση στα οικονομικά, προσιτά οικονομικός δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και λιγότερο δυσκίνητες ε, ρυθμίσεις. Επίσης αποφυγή αλληλεπικάλυψη των ε, εθνικών ερευνητικών συστημάτων. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πιο εύκολο για τους ε, φορείς καινοτομία και τους ερευνητέ να εργάζονται ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Αυτό μέχρι στιγμής δεν είναι τόσο εύκολο. Επίσης πιστεύουμε ότι το ειδικευμένο ε, εργατικό δυναμικό είναι πολύ σημαντικό για μια βιώσιμη και καινοτόμο οικονομία και είναι μια, ένα ακόμα από τα σκέλη της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Υπάρχει και στόχος απασχόλησης στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες ε, και να ομοιογενοποιήσουμε κάπως ε, τις δεξιότητες σε σχέση μεγαλύτερη ε, μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης, κάτι που δεν έχουμε επιτύχει. Και η βιομηχανία θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο, όχι μόνο υπηρεσίε, αλλά η βιομηχανία πρέπει επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και αν δείτε κάποιες χώρες ε, που έχουν καλές επιδόσεις θα δείτε ότι η ισχύ τους βασίζεται στο βιομηχανικό τομέα κατά κύριο λόγο. Στο μέτωπο αυτό η στρατηγική αποσκοπεί ε, στην πρόθεση της απασχόλησης και στη διατήρηση διαφοροποιημένης και ισχυρής βιομηχανικής βάσης Εν τέλει, μια δυο, μια ε, για τις ε, γενικότερες παγκόσμιες προοπτικές. Ε, υποστηρίζουμε το έργο του G20 στο μέτωπο αυτό γύρω από την ανάπτυξη, πρωτοβουλία ανάπτυξης της, του G20 και σχέδιο δράσης. Όλα αυτά θα πρέπει να άλληλο υποστηρίζονται με στόχο να βοηθήσουμε αυτούς που θα πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις αλλά και αυτούς που θα πρέπει να τις υλοποιήσουν ώστε να έχουμε πράγματι εξελίξεις και πρόοδο. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι, ολοκληρώνοντας, ότι είναι σαφές ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα σχεδιαγραφούμε τι προτεραιότητές μας κατά κάποιο τρόπο με βάση τις αναλύσεις μας και δεύτερον προσπαθούμε να ορίσουμε το πλαίσιο ώστε να βοηθήσουμε ίσως και να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις σε επίπεδο πολιτικής δεν θέλουμε βέβαια ε, να, θέλουμε να διατηρήσουμε την ακαιρότητα της όλης αυτής ε, διαδικασίας και θέλουμε όλα τα επίπεδα, εθνικά, ε, Εθνικό Κοινοβούλιο, Κοινωνική Εταίρη, Ευρωπαϊκό επίπεδο επίσης, πάλι Κοινωνική Εταίρη. Όλοι θέλουμε να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή. Δεν θέλουμε να είναι κάτω που κάνουν οι δημόσιε διοικήσει. Δεν θέλουμε να είναι ένα πρόγραμμα εργασίας. Ένα πρόγραμμα το οποίο το μαγειρεύουν οι υπάλληλοι της Κομισιόν ή οι εθνικοί αξιωματούχοι. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό οι προτεραιότητες αυτές να είναι κοινέ, πραγματικά κοινέ. Και οπουδήποτε βρισκόμαστε, αυτό το τονίζουμε και σκοπός μας είναι να βάλουμε μα μας τις δυνάμεις ώστε να γίνουν ε, πράξη οι πρωτοβουλίες μας. Καλές είναι οι πρωτοβουλίες, αλλά αυτό που θέλουμε είναι αποτελέσματα και τον Ιούνιο θέλουμε να δούμε τι πολιτικές έχουν τα κράτη-μέλη και να δούμε μετά και να πούμε όχι δεν, είναι, δεν αρκεί ή αρκεί, είναι στο πορεία κτλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή αυτή που κάνατε συζήτηση. Δύο συντονιστές λείπουν, ο Ότμαρ Κάρας ασθενή και η Περβάνος Μπερές λαμβάνει μέρος σε ένα κοινωνικό φόρουμ, οπότε δεν είναι εδώ παρούσα. Οπότε θα ζητήσουμε μια τοποθέτηση από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν ξέρω ποιος θέλει να μιλήσει. Ντανούτα. question, e Ναι, Κάποιος είναι εδώ από το ΕΛ και η απάντηση είναι ναι. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι και να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε πως οι κυβερνήσεις αύξησαν τις δαπάνες για να αντιμετωπίσουν την κρίση, γι' αυτό βρέθηκαν εδώ που βρέθηκαν. Και τώρα πρέπει να κάνουν οικονομίες. Είναι λίγο απλοποιημένη αυτή η δήλωση. Γιατί δεν ήταν μόνο θέμα οικονομικού κύκλου ε, που είναι φυσικό η κυβέρνηση να ξοδεύει παραπάνω όταν υπάρχει συρρήκνωση, αλλά υπάρχει, υπήρξε, υπήρξαν αυξημένε δαπάνε που δημιούργησαν προβλήματα, όχι λόγω της κρίσης ε, σε καιρού ε, ύφεση, αλλά λόγω των προβλημάτων στον τραπεζικό τομέα τα μεγαλύτερα προβλήματα νομίζω σχετίζονταν όχι με την οικονομική κατάσταση αλλά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οπότε χρειαζόμαστε εξαιρετικούς ή ειδικού κανόνες ή μέσα για να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση. Όταν ε, μιλάμε για το δημόσιο χρέος. Γιατί μόνο με απλή ανάκαμψη και ανάπτυξη δεν θα μπορέσουν ε, τα κράτη-μέλη να επανέλθουν στα συνήθη και να αναλάβουν το ρόλο τους ε, ως ε, πάροχοι κρατικής χρηματοδότησης. Οπότε πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερη προσοχή στο θέμα αυτό της κατάστασης των προπολογισμών και να είμαστε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά το πώς θα γίνει η εξοικονόμηση και πώς θα μπορέσουμε να έχει ξανά το κράτος ε, τον ρόλο του όσον αφορά τις δημοσίες δαπάνες. Οπότε εδώ η Ευρώπη 2020 τα βάζει όλα αυτά κατά μέρο και κάνει μια διαφορετική συζήτηση για την οικονομική διακυβέρνηση και όχι ε, για το θέμα το οποίο επίσης ισχύει εδώ πέρα, δηλαδή η εθνική προπολογισμή, στο πλαίσιο του πώς θα βγούμε από την κρίση μέσω χρηματοδότησης. Οπότε οι οικονομίες ε, και το πώς θα γίνουν είναι κάτι ε, το οποίο αξίζει πολύ περισσότερης προσοχής για το πώς θα βγούμε από την κρίση και μετά Μιλάτε για το, ελκυστικό, για το πώς θα προσελκύσουμε ιδιωτικό κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη. Υπάρχει μια απλή συνταγή και είναι τα ομόλογα έργων. Και μετά θα υπάρχουν κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ξέρουμε πόσο δύσκολο ήταν βεβαίως πάντα για τις Ευρώπη να δημιουργήσει τέτοια κεφάλαια. Και δεν είναι σαφές ε, γιατί τη στιγμή που υπάρχει μια απομάκρυνση από την ανάληψη κινδύνου θα εμφανιστεί τέτοιο κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια πραγματική αλλαγή δηλαδή όσον αφορά την πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση όταν μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων και των τραπεζών δεν βλέπουμε κάποια συνεργασία και πρόσβαση σε χρηματοδότηση και θα λύσουν ε, πράγματι όλα τα ζητήματα χρηματοδότηση επενδύσεων τα ομόλογα έργων. Επίσης εκπλήσωμαι από το ότι δεν αναφέρεται καθόλου ο προπολογισμό τη Ένωσης σε όλη αυτή τη συζήτηση περί χρηματοδότηση ανάπτυξη. Οπότε μπορείτε να μας πείτε σε ποιο βαθμό αυτές οι εύκολες από ό,τι φαίνεται συνταγές είναι ρεαλιστικές. Και πώς ε, θεωρείτε ότι οι εθνικοί προπολογισμοί μπορούν να υποστηρίξουν τον καταλητικό ρόλο που έχουν Όταν, πότε δηλαδή θα ανακάμψει αυτή του τους η λειτουργία. Ε, Ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες και ερωτήσεις και τα χρήσιμα σχόλια. Ήταν περισσότερο σχόλια αυτά που είπατε πατά, παρά ερωτήσεις. Σας είπα στην αρχή ότι δεν θα μιλήσω για την δημοσιονομική εξυγίανση. Η προσέγγιση της Κομισιόν είναι μία πλήρης, μία εμπεριστατωμένη προσέγγιση. Είναι εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, χρηματοπιστωτικό τομέας και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη. Εσείς στα σχολιά σας καλύψατε και τα τρία. Η δημοσιονομική εξυγίανση γίνεται με πολλούς τρόπους. Εξαρτάται από τη χώρα. Τι πορεία είχαν, γιατί φτάσαν σε αυτό το επίπεδο ελλείμματο κτλ. Αλλά πιστεύουμε ότι αυτή η εξυγίανση είναι σημαντική, γιατί αλλιώ οι χώρε δεν θα μπορέσουν να έχουν κανένα περιθώριο λιγμού στο προπολογισμό του και δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν αυτό που πρέπει να χρηματοδοτήσουν. Τώρα, πώ θα κινηθεί κάθε χώρα εξαρτάται. Έχουμε τι ακραίε περιπτώσει όπου κάποιε χώρε υφίστανται κάποια προγράμματα και έχουν εξωτερική χρηματοδότηση. Υπάρχουν χώρε όμω που δεν το χρειάζονται έχουν συμφωνήσει ε, για μια πολυετή περίοδο εξυγίασης. Παράλληλα θα πρέπει να κρατήσουν ε, ένα επίπεδο βιωσιμότητας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που εμποδίζει τη χώρα για να κάνει τις σωστέ δαπάνες ε, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη. Τώρα πώς θα γίνει η εξυγίαση. εμείς τονίζουμε ότι κάθε χώρα θα πρέπει να δει τη σύνθεση, από πού θα προέλθει αυτή η εξυγίανση. Είναι, έχουν σημασία οι λεπτομέρειες. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο το έλλειμμα. Πρέπει να κοιτάμε τις δαπάνες, τι γίνεται με τους φόρους, ποια είναι η καλύτερη σύνθεση του μείγματος της εξυγίανσης. Γιατί ε, η επίπτωση στην πραγματική οικονομία διαφέρει ανάλογα με το μείγμα της εξυγίανσης. Ξέρετε τη συνήθεια διαδικασία που ακολουθούμε με τις χώρες. Σε πρώτη φάση κάνουμε μια αξιολόγηση του προγράμματος σταθερότητας και σύγκλησης. Θα κοιτάξουμε τους προπολογισμούς, ε, τις προτάσεις προπολογισμού για το 2012 και θα δούμε αν συνάδουν με την προσπάθεια εξυγίανσης. Στο σημερινό πακέτο το οποίο συζητά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υπάρχουν πολλές προτάσεις για να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο χρέος και στην εποπτεία του δημοσιονομικού άξονας, πολύ περισσότερο από την παλιά και του φορολογικού στοιχείου. Αυτά περί Τώρα, για τα ομόλογα έργων. Φυσικά από μόνο δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα της κρίσης. Ωραίο θα ήταν, θαυμάσιο, αν μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο με αυτά τα ομόλογα. Είναι μία από τις δυνατότητε που έχουμε που θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε για να τη χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο που μπορεί να ελκύσει και άλλες επενδύσεις ούτως ώστε να υπάρξουν αυτές οι διασυνοριακές επενδύσεις. Είμαστε σε φάση δρομολόγησης ακόμα. Αν δεν απατώμε, πολύ σύντομα θα γίνει και μια πρόταση όχι ακριβώ πρόταση, αλλά πώ θα το κάνουμε. Μετά θα γίνουν διαβουλευσει και μετά θα γίνει η πραγματική πρόταση για αυτά τα ομόλογα έργων και το πώ μπορούν να εφαρμοστούν. Τώρα για τον τραπεζικό τομέα. Ε, εδώ συμβαίνουν πολλά πράγματα στον τραπεζικό τομέα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει το νομοθετικό πακέτο για το χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο ετοιμάστηκε πέρυσι. Όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν τώρα στη θέση τους. Ε, το είδος της χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Θα κάνουμε και άλλες ε, δοκιμές ε, αντίστασης. Δοκιμές κόπωσης στις τράπεζες. Και η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα όλο και περισσότερο αποτελεί τμήμα των κοινοτικών συστάσεων. Το έχουμε στο μυαλό μας για χώρες υποπρογράμματα, αλλά και για αυτές που δεν υφίστανται κανένα πρόγραμμα. Είναι τμήμα, ας πούμε, των υποχρεώσεων που έχουν οι χώρες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχουν ένα πρόγραμμα, δηλαδή, για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Το τελευταίο στοιχείο είναι η χρηματική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δύο μηχανισμοί που αναπτύσσονται για την Ιρλανδία και την Ελλάδα. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε έναν μόνιμο μηχανισμό τώρα. Ε, μέχρι στιγμής έχουμε αυτό τον, ε, το μέσο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ε, το Μάρτιο θα αποφασίσουμε. Όμως... Κανονικά πρέπει να μιλήσει η Κίνγκα Γκένσου, αλλά θα ήθελα να αλλάξουμε αν θέλετε γιατί πρέπει ο Λεσμίτ να πάει αλλού σε 4. Α, και εσεί θα πάτε σε άλλη συνεδρίαση. Τότε θα μιλήσετε και οι δύο. Θα μιλήσετε, κάντε την ερωτήση σας και θα απαντήσετε εσείς μαζί. Με συγχωρείτε, αλλά ξέρετε έχουμε πτήσεις όλοι μας να προλάβουμε. Κατά βάση συμφωνώ με αρκετά από αυτά τα οποία είπατε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια επίσης. Όταν μιλάμε για εξυγίανση των προπολογισμών, από τη μία συμφωνούμε πως είναι απολύτως απαραίτητη, από την άλλη συμφωνώ πως μπορούμε να απλοποιήσουμε την... Ε, απλοποιούμε έτσι την κατάσταση, γιατί βλέπετε τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Οπότε αν έχουμε κάποια ανάκαμψη χωρίς ε, ε, βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας, ε, τότε νομίζω πως ε, στο μακροεπίπεδο θα έχουμε καλύτερα δεδομένα και η κατάσταση θα βελτιώνεται, αλλά όχι στο, στο μικροεπίπεδο. Και βλέπουμε ένα χάσμα όσον αφορά την εδαφική συνοχή, κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη και πρέπει να, το, να τα αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε ειδικά προγράμματα για ειδικέ ομάδες, ε, άνεργους νέου, ε, άνεργους ε, μακροπρόθεσμα και ανέργους που ανήκουν σε ευπαθεί ομάδε. Είναι μεγάλος ο κατάλογος. Επίσης, μιλάμε για την πράσινη ανάπτυξη, αλλά πρέπει να ορίσουμε πως ε, να διευκρινίσουμε πως χρειάζεται επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη, στο να προετοιμάσουμε τον κόσμο στο να περάσουμε από μια βιομηχανική γεωργία σε μια πράσινη γεωργία για να υπάρξει μια σωστή μετάβαση σε αυτή τη βιομηχανία και χρειάζεται βέβαια ο απαραίτητος μηχανισμός. Χρειάζεται επίσης μια ολοκληρωμένη τέτοια περιοχή στην Ευρώπη. Οπότε εμεί θα θέλαμε να τονίσουμε πως στρατηγική του 2020 χωρίς πόρους και περισσότερο συντονισμό μεταξύ εθνικού και κοινοτικού επίπεδου χρηματοδότησης παραμένει στο επίπεδο των ε, ευχολογίων και τη χρηματοδότηση να αναφέρατε, τα ευρωομόλογα, εγώ θα ανέφερα και την εισαγωγή ενός φόρου στις ε, χρηματοοικονομικής συναλλαγής γιατί λεφτά υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς ε, θα μπορέσουμε να βρούμε ένα μηχανισμό για να διοχετεύσουμε αυτά τα λεφτά στον παραγωγικό τομέα και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Για να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τα κονδυλία Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Το έγγραφο αυτό να το δούμε μπορούμε να πούμε πως είναι πολύ φιλόδοξο και βεβαίως ίσως στο τέλος όλα πάνε καλά αλλά εάν δείτε τα διαγράμματα και το κείμενο είναι θλιβερή αυτή η ιστορία που περιγράφεται για την Ευρώπη και για την ευημερία της Ευρώπης. Το ποσοστό φτώχειας, ποσοστό ανεργίας κτλ. Και Κοιτώντας την εισαγωγή σας εδώ πέρα, λέει πως η Κομισιόν σκοπεύει να διερευνήσει με τα κράτη-μέλη ε, το τι θα κάνει και το πώς ε, θα καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κτλ. Και αφήνοντας το χρήμα κατά μέρος, τι, τι σκοπεύετε να κάνετε. Εγώ αν ήμουν υπουργό και το κοίταγα αυτό το έγγραφο, δεν θα ήμουν και πολύ ικανοποιημένο. Εάν δείτε τους πίνακες, βλέπετε πως η Ολλανδία δεν έχει στόχους καθόλου. Δεν αναφέρονται κάποια πράγματα. Τουλάχιστον ε, όχι στο έγγραφο στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης. Και σε κάποιους από τους στόχους υπάρχουν λιγότερα νούμερα. Δεν ξέρω, ίσως λίγες μόνο χώρες μπορούν να πούν ποιοι είναι οι στόχοι τους. Πρώτα απ' όλα νομίζω πως χρειαζόμαστε στόχους και εσείς χρειάζεστε, στό, χρειάζεστε στόχους εάν είναι να βοηθήσετε τις ε, χώρες ε, στο να εισαγάγουν μεταρρυθμίσεις. Τι, τι άποψη έχετε. Είναι τι, το, το εφικτό. Είναι, δυνα, είναι να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Και Ποιε είναι οι διαφορέ από την στρατηγική τη Λισαβόνα, τι άποψη έχετε για τη γαλλογερμανική πρωτοβουλία, είναι κάτι θετικό, αρνητικό ή, είναι κάτι που μπορεί να ευθυγραμμιστεί με αυτά τα οποία κάνετε εσεί ή θα συγκρουστεί. Θα υπάρξουν τριβέ. Και εγώ ειλικρινά ελπίζω για το καλύτερο γιατί μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης. Και όταν διαβάζω πως η φτώχεια στην Πορτογαλία ε, όταν ήμασταν εκεί πριν από λίγες εβδομάδες ε, εκπλήσωμε που συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη σήμερα ε, είναι τη 2011 Ίσως να είναι χαζή ερώτηση αλλά μου την έκαναν στην πατρίδα μου και δεν μπορούσα να απαντήσω. Πού είναι η μείωση της φτώχειας, γιατί την αναφέρετε εδώ Τι σημαίνει μείωση της φτώχειας και η γραμμή της φτώχειας στην Ευρώπη Φαντάζομαι πως δεν είναι το ίδιο το όριο στη Σουηδία και στην Πορτογαλία. Ποιο είναι το όριο της στόχιας, είναι 60% του μέσου μισθού, τι είναι. Εδώ πέρα λέει κάποια πράγματα στα σχόλια, αλλά δεν ξέρω, μπορείτε να μου βοηθήσετε για να απαντήσω και εγώ στους ψηφοφόρους μου την επόμενη φορά. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μάλλον δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να σας πω αυτά που ξέρω και αυτό το οποίο κατάλαβα ως ερώτηση και την άποψη της Κομισιόν για το σχόλιο σας για την ανάκαμψη και το ότι υπάρχει στο μακροεπίπεδο αλλά όχι στα άλλα επίπεδα. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ πως βασικά είναι στοιχείο σύνθεσης ε, των εθνικών προϋπολογισμών, δηλαδή σε ποιο βαθμό διαχέεται η ανάκαμψη στο εθνικό επίπεδο και η προσπάθεια ε, που γίνεται τώρα διανέμεται και πώς διανέμεται. Και νομίζω πως ε, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το δει κανεί μόνο εάν δει του εθνικού προπολογισμού. Γιατί εκεί πέρα βλέπουμε ποιο καταβάλει προσπάθειε και ποιο ε, δεν καταβάλει. Βλέπετε πού πάνε τα λεφτά, από πού προέρχονται οι φόροι και φαίνεται αυτό πάρα πολύ καλά. Αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα γιατί είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Αλλά τουλάχιστον για εμάς ε, στην Κομισιόν εμείς δεν είμαστε σε θέση να μπούμε σε αυτά, αλλά είμαστε σε θέση να πούμε πως ε, η κατανομή της προσαρμογής είναι σημαντική και πρέπει να ληφθεί υπόψη αν θέλουμε να γίνει προσαρμογή, αλλιώς δεν θα είναι εφικτή γιατί δεν θα είναι αποδεκτή και ταυτόχρονα ε, έτσι πρέπει να σκεφτούμε το τι θα γίνει μετά την προσαρμογή, το πώς θα έχει η κατάσταση αλλά αυτό είναι πολύ πολιτικό ζήτημα και αν δείτε προπολογισμού διαφορετικών χωρών βλέπετε διαφορετική κατανομή. Είναι ένα στοιχείο αυτό λοιπόν. Για τα διάφορα πράγματα που είπατε για τις πολιτικές που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την πράσινη ανάπτυξη και την αύξηση των εσόδων, στο μέτωπο αυτό αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε το τι θα μπορούσε να γίνει. Τίποτα δεν έχει αποκλειστεί, τα μελετάμε, άλλα είναι σε το τεχνικό επίπεδο, άλλα είναι στα έγγραφα της Κομισιόν, αλλά σαφώς όλα αυτά τα ζητήματα, ε, το ξέρω, αν και είναι στο τεχνικό επίπεδο, π.χ. για την φορολόγηση διαφόρων ε, χρηματοοικονομικών συναλλαγών αρχίζουμε και μελετάμε μοντέλα για να δούμε τι αντίκτυπο θα έχουν. Οπότε υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην το βλέπετε αυτή τη στιγμή στα έγγραφα της Κομισιόν. Υπάρχουν. Για την ερώτησή σας για το πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα συμβούν όλα αυτά. Αυτό είναι το θέμα της εφαρμογής. Το πώς από το ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή όλων αυτών των δεσμεύσεων ή συστάσεων που, σοπιές συμφωνούν οι χώρες ή συστάσεων που κάνει η Ένωση στις χώρες. Νομίζω πως από αυτό το πρίσμα, το, αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με το νομοθετικό πακέτο που είναι τώρα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι να αυξήσουμε τις δυνατότητες εφαρμογής και επιβολής, δηλαδή να υπάρξει άλλο ένα στρώμα πίεσης στις ε, χώρες όσον αφορά τις συστάσεις που τους γίνονται στο επίπεδο της Ένωσης και όσο περισσότερο μπαίνει αυτό στην εθνική συζήτηση τόσο το καλύτερο γιατί τότε η πίεση θα έρθει και από τα εθνικά κοινοβούλια κτλ. Οπότε δεν θα είναι μόνο ευρωπαϊκή. Οπότε η επιβολή είναι ένα κίνδυνο. Έχουμε ε, εργαλεία, αλλά είναι πάντα ένα κίνδυνο. Δεν σημαίνει επειδή έχουμε στόχους ε, και ε, μέτρα σύγκρισης ότι θα το επιτύχουμε. Αυτά είναι εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν. Όλα αυτά συμπληρώνουν τις ε, πολιτικές, αλλά νομίζω πως έχουμε τώρα κάποιες προτάσεις ε, επιτάπητος που μπορούν να ενισχύσουν νομίζω σημαντικά το κομμάτι της ε, επιβολής. Και επίσης ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να είμαστε εστιασμένοι είναι ακριβώς για να υπάρχει αυτή η καλύτερη επιβολή και εφαρμογή. Πάντα υπάρχει ε, αυτός ο διχασμός γιατί κάποια τονίζουμε και μετά μας λένε «Ε, δεν τονίσατε τα άλλα κτλ. Αλλά όπως είπα και στην αρχή με 10 προτεραιότητες ή με 3 συστάσεις πολιτικής ε, μπορούμε να πούμε πως το επόμενο έτος τα κάνατε ή δεν τα κάνατε και ποιο ήταν το αποτέλεσμα όσον αφορά τους δείκτες. Και εφόσον το κάνουμε αυτό κάθε χρόνο μπορούμε να εστιάσουμε στα σημαντικά κάθε φορά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αλλά βεβαίως Χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Τώρα για τη γαλλογερμανική πρωτοβουλία. Ε, δεν ξέρω, κοίταξτε, εγώ το λέω... Το λέω όπως το λέτε κι εσείς, έτσι, γιατί είναι θέμα το πιανού είναι η πρωτοβουλία. Από αυτά τα οποία ξέρουμε, γιατί από ό,τι ξέρετε δεν υπάρχουν γραπτά και τίποτα, όλα αυτά αλλάζουν. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς ότι είναι η πρωτοβουλία είναι πως ε, εάν αναπτυχθεί σωστά θα μπορέσει να αποτελέσει ένα ακόμα στρώμα επιβολής. Δηλαδή αν υπάρξει ακόμη μια δέσμευση στο επίπεδο αρχηγών κρατών σε κάποιες από αυτές τις πολιτικές προτεραιότητες και πούν παραδείγματο χάρη οι χώρε Ευρωζώνη ε, θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα, να λαμβάνουν αυτή τη δέσμευση κτλ. Οι υπόλοιπε χώρε μπορεί άμα θέλουν και αυτέ. Αυτή θα είναι μια επιπλέον πίεση. Έτσι βλέπω εγώ την συμβατότητα ε, στο πλαίσιο της πολιτικής. Όσον αφορά την ουσία, νομίζω πως ε, όλα αυτά πάνε προς την ίδια κατεύθυνση αλλά οι ιδέες που ακούσαμε ούτως ή άλλως θα εξελιχθούν, γιατί από ό,τι κατάλαβα κάποιες ιδέες ε, αναφέρθηκαν, ε, που αναφέρθηκαν ε, από τη Γερμανίδα Καγκελάριο δεν έγιναν τόσο καλά δεκτές. Οπότε τα πράγματα εξελίσσονται και ίσως να μην γίνουν όλα αυτά δεκτά από όλες τις χώρες. So, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τη σημερινή συζήτηση που μας παρέχει και τις πληροφορίες. Θα με συγχωρέσει όμως να πω ότι συγκρατώντας αυτό που είπε ότι όχι μόνο οι πολίτες αλλά και εμείς οι ευρωβουλευτές ακούγοντας στρατηγική 2020, οικονομική διακυβέρνηση, συμφωνανταγωνιστικότητα και διάφορα άλλα τέτοια βρισκόμαστε, ας το πω έτσι, σε μια σύγχυση. Τι είναι όλα αυτά, πώς συνδέονται, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, <laughs> ποιο θα εφαρμοστεί τελικά. Και ξέρετε αυτό με μια ρητορία, ε, με ωραία πράγματα μπορεί να το ξεπεράσεις. Αλλά κατά τη γνώμη μου, και εδώ είναι το σχόλιο και δεν αφορά προσωπικά την Επίτροπο που καταβάλει προσπάθειες να μας τα ξεκαθαρίσει, εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα, είναι μαζί με την κρίση την οικονομική και την κοινωνική έχουμε κρίση πολιτικής και κρίση πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέρος αυτής της κρίσης είναι και η Κομισιόν. Και θα σας πω γιατί. Όλο αυτό το κείμενο της στρατηγικής ε 2020 ε, ε, ε, έχει τη σκουριά, τη σκουριά της στρατηγικής της Λισαβόνας. Έχετε χάσει την αίσθηση της πραγματικότητας, της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και των προβλημάτων. Θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα για να μην σας τρώω πολύ το χρόνο αυτά που λέτε πρώτον είναι αλληλοσυγκρόμενα και δεύτερο, όπως θα σας αναφέρω παράδειγμα, υπερβαίνουν και παραβιάζουν τη συνθήκη. Τη συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυτά που λέτε. Πρώτο παράδειγμα. Σφιχτή δημοσιονομική πολιτική και κυρίως εξυγίανση των δημοσιονομικών διαφόρων χωρών και αντιμετώπιση του προβλήματος της ανάπτυξης και της απασχόλησης δεν έχω δει πουθενά. Σας αναφέρω πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα από τη χώρα μου την Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε καθεστώς μνημονίου, βρισκόμαστε σε καθεστώς να μαζέψουμε τα δημοσιονομικά μας γιατί το ξεχυλώσαμε, σύμφωνοι, και τώρα μιλάμε πώς θα μαζέψουμε όλα αυτά και ταυτόχρονα ακούγεται και το θέμα της ανάπτυξης και της αντιμετώπιση της απασχόλησης. Πράγματι, από τα κοινοτικά ταμεία δίδονται χρήματα τέσσερα προγράμματα για την αντιμετώπιση τη απασχόληση. Έτσι. Νέε θέσει εργασία να χρηματοδοτηθούν, να επανεκπαιδευτούν οι άνεργοι. Το πρόβλημα όμω πού είναι. Η απορροφητικότητα αυτών των κονδυλίων από την πλευρά τη ελληνική κυβέρνηση είναι χαμηλή. Όχι από γραφειοκρατικέ αγκυλώσει, αλλά γιατί το εθνικό μερίδιο στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δεν μπορεί να δοθεί. Διότι έχουμε περικοπή των δημοσίων δαπανών. Επομένω, έχουμε μια σύγκρουση. Πώ θα υπάρξει ας πούμε ανάπτυξη και αντιμετώπιση του προβλήματος τη απασχόληση στην Ελλάδα που είναι μεγάλο όταν η μία προτεραιότητα και η μία κατεύθυνση συγκρούεται. Και σε αυτήν επιμένετε σε μία από τι δράσει σα. Λέτε εδώ στι 10 δράσει, έχω μπροστά το κείμενο, ότι θα θέλουμε να επανέλθουν οι άνεργοι στην απασχόληση. Και πάω στο δεύτερο παράδειγμα. Ανάμεσα στι 10 δράσει που αναφέρετε, μιλάτε για τη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Σας ερωτώ τώρα λοιπόν. Είναι δυνατόν αφού το άρθρο 153 λέει ότι η Ένωση δρά επικουρικά και σέβεται τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης της κάθε χώρας και δεν επηρεάζει την πολιτική τους ούτως ώστε να μην χαθεί η αισθητά οικονομική ισορροπία εσείς να απαιτείτε όχι επικουρικά όπως προέβουν οι συνθήκες αλλά με την έννοια μιας καθολικής επιβολής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού των συνταξιδοτικών συστημάτων αφού είναι μία από τις δράσεις να απαιτείται η παρέμβαση να παραβιάζει την ε, εθνική δυνατότητα και να παραβιάζει τις συνθήκες και το άρθρο 153 τις συνθήκες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν συγκρούεται. Πώς θα, το, πώς θα πραγματοποιηθεί, τι θα κυριαρχήσει. Και από όσο ξέρω το άρθρο 153 δεν το έχετε για μεταρρύθμιση, για αλλαγή, έχουμε μόνο το 136. Κατόπιν τούτου θα σας έλεγα για να μην σας στεναχωρήσω περισσότερο, ωραία είναι αυτά, ωραία μας τα λέτε, αλλά νομίζω και δεν γελώ τώρα, γελώ έτσι χαριτολογώντας ότι τα αποτελέσματα θα είναι κάτω από τις προσδοκίες ήδη φαίνονται, ακόμα και κάτω από αυτές τις ψευδεστήσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας που έλεγε για πιο ανταγωνιστική οικονομία και για πλήρη απασχόληση στην Ευρώπη. Θα έχουμε μάλλον επιδείνωση και στους δύο δείχτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια ένταση. Κάθε φορά που πρέπει να προβούμε σε δημοσιονομική εξυγίανση υπάρχει ένα αντιστάθμισμα. Δηλαδή υπάρχουν εντάσεις. Μ' Τώρα, πώς θα επιλύσουμε τις εντάσεις αυτές. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πει πολλά. Είναι... Μ' ακούτε, δεν μ' ακούτε. Μ' ακούτε εντάξει, ε, κύριε Χουντή, ωραία. Είναι φυσιολογικές αυτές οι εντάσεις όταν θέλουμε να κάνουμε εξυγίανση. όταν δεν έχουμε... Προφανώς δεν έχουμε όλα τα λεφτά για να πληρώσουμε τα πάντα. Πώς θα επιληθεί το πρόβλημα αυτό των εντάσεων είναι θέμα πολιτικών επιλογών. Ε, εξαρτάται όμως και από τα χάσματα που έχουμε. Αν σκεφτούμε την κατάσταση στην Ελλάδα τώρα. Είναι από τις πιο δύσκολες. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες ε, αντιμετώπισαν αντίστοιχες καταστάσεις το 2008 και 2009 είχαμε την Ουγγαρία και τη Λετωνία, κυρίως αυτές τις χώρες. Αλλά κάποια στιγμή κανένας δεν θέλει να αγοράσει δημόσιο χρέος. Και όταν κανένας δεν θέλει να αγοράσει δημόσιο χρέος, είσαι κολλημένος στον τοίχο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να επιλέξεις αν θα έχει ε, επιδόματα για την ανεργία, αν θα έχει δαπάνε για την καινοτομία, δεν μπορεί να πληρώσει καν του μισθού. Αυτό μην το ξεχνάμε. Αυτό είναι το σημείο αφετηρίας. Τώρα, για να μην αναφερθώ στους λόγους, ε, δεν νομίζω ότι είναι ο σκοπός της συζήτησής να κάνουμε αυτή την ανάλυση γιατί φτάσαμε εδώ, αλλά να έχουμε υπόψη μας αυτό το σημείο αφετηρίας, γιατί αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση που θα αντιμετωπίσει ειδικά η Ελλάδα θα είναι πολύ δύσκολη. Εδώ θα πρέπει να γίνουν επιλογές. Και ευτυχώς ή δυστυχώς ήμουν επικεφαλής του προγράμματος ε, των χωρών που ανέφερα, δηλαδή Ουγγαρία και Λετωνία, όχι για την Ελλάδα, δεν ήμουν υπεύθυνη και ξέρω τι κάναμε. Ε, είδαμε γραμμή προ γραμμή τον προϋπολογισμό και αυτό είναι πολύ επώδυνο. Μαζί με την κυβέρνηση ψάξαμε κάθε δημοσιονομική γραμμή, συζητήσαμε με τους κοινωνικούς εταίρους κάθε γραμμή του προϋπολογισμού, κάθε δαπάνη, κάθε φόρο και συμφωνήσαμε με τις εθνικές αρχές τι θα κάνουν ούτω ώστε να τις βοηθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρξουν δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δάνεια που δεν μπορούσαν να, πάνε, να πάρουν από αλλού. Τώρα, πάλι πρέπει να κάνεις εδώ επιλογές. Παραδείγματο χάρη, συλλογή φόρων. Έτσι. Ξέρω ότι το επίπεδο συλλογής φόρων στο χαρτί με, την, τα πραγματικότητα έσοδα από τη φορολογία απέχουν πάρα πολύ. Όταν κάνει τους υπολογισμούς αυτό, αυτή η διαφορά είναι τεράστια. Αν όμως ε, λειτουργεί σωστά και σε αυτό το επίπεδο θα μειώσει τις εντάσεις. Καταλαβαίνω ότι δεν είμαι πολύ ακριβής τώρα, αλλά καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ε, είναι πολύ δύσκολη η συγκυρία, πολύ δύσκολη αυτή η προσπάθεια, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Επίση, δεύτερο στοιχείο, ω προ τι δαπάνε, Θα πρέπει τα ευρωπαϊκά κονδύλια να πάνε στη σωστή μεριά. Είναι πολύ σημαντικό ούτω ή άλλω αυτό, αλλά σε εποχέ κρίση είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το αν, α πούμε, τα κονδύλια από το Ταμείο Συνοχή, ε, τα διαφορετικά ταμεία κτλ., ακόμα και τα λεφτά για την έρευνα, έχει σημασία που πάνε πρέπει να το ψάχνουμε πολύ λεπτομερώς, ούτω ώστε κάθε ε, ευρώ να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα για το συνταξιοδοτικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ε, αντίφαση και σύγκρουση. Γιατί αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και όχι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το κάνουμε από κοινού με τα κράτη-μέλη, ό,τι κάνουμε. Δουλέψαμε πάρα πολύ εδώ και 10 χρόνια για τη βιωσιμότητα και μια, μια ανάλυση βιώσιμη. Και όλοι συμφωνούμε με το συμπέρασμα ότι τα περισσότερα συνταξιδοτικά συστήματα δεν είναι βιώσιμα λόγω των δημογραφικών τάσεων. Και επομένως το συμπέρασμα είναι ότι τα περισσότερα συστήματα πρέπει να αλλάξουν κατά ανάγκη. Εμείς δεν μπαίνουμε στο πώς θα αλλάξετε εσείς τα συστήματά σας πόσο τμήμα του δεύτερου πυλώνα θα πρέπει να είναι ιδιωτικό. Δεν μπαίνουμε σε τέτοια, τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτά είναι θέματα εθνικά. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας, θέμα επιλογών των κυβέρνησης. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να γίνουν κάποια βήματα και τα βήματα αυτά είναι αναπόφευκτα, δυστυχώς. Να παρέμβω. Γιατί αυτή η προσπάθεια εξυγίανσης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Στην Ουγγαρία, ας πούμε. Θεωρείτε ότι το, το εθνικό σταξιδοτικό σύστημα είναι σωστό. Ή παραδείγματο χάρη ότι η εξυγίαση του φορολογικού συστήματος ή του δημοσιονομικού συστήματος πηγαίνει προς την ορθή κατεύθυνση. Το σταξιδοτικό, ας πούμε, είναι βιώσιμο στην Ουγγαρία. Φοβούμαι ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί θα έπρεπε να γνωρίζω ακριβώς τι έχει γίνει. Δεν το γνωρίζω, αλλά θα μπορούσα να σας απαντήσω σε μεταγενέστερο στάδιο. Λυπούμε. Δεν ξέρω ακριβώ ε, τι έχει γίνει. Έχει γίνει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο προπολογισμό, είναι ένα ξεχωριστό προπολογισμό. Δεν, δεν γνωρίζω. Λυπούμε. Κυρία Ολμάια. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως η συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα γιατί οι παρατηρήσεις ε, της εισηγήτριας εδώ πέρα και κάποια από αυτά τα οποία διαβάζω εδώ πέρα στην έκθεση λένε πως κάποια από τα προβλήματα αυτά προϋπήρχαν της κρίσεις και δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά και δεν οφείλονται αποκλειστικά στην ε, οικονομική κρίση. Και εκεί πέρα ανήκει το ζήτημα της υπερβολικής ε, χρέωσης και δαπανών ε, χρημάτων που δεν υπήρχαν. Και φοβάμαι πως ε, τελικά αυτά θα επανέλθουν με κάποια καθυστέρηση. Εντός της Ένωσης υπάρχουν διαφορετικά ε, κράτη-μέλη, ανέφεραν οι συνάδελφοι την Ελλάδα. Η Ελλάδα πράγματι προχώρησε πραγματικά πάρα πολύ ε, μακριά γιατί de facto ήταν ε, στα, όρια της χρεοκοπίας αν δεν υπήρχε ε, η βοήθεια από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως βγάλε τα απαραίτητα συμπεράσματα και κινήθηκε λόγος. Το θέμα λοιπόν είναι πως τα συμπεράσματα από την Ελλάδα είναι σχετικώς προφανή αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε το τι θα γίνει σε περίπτωση σαν την Ελλάδα. Δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, μπορούσε να είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα κράτη-μέλη. Λοιπόν, πόσο επιτυχείς είμαστε στο να δημιουργήσουμε μεσαίες επιχειρήσεις που θα ε, έχουν προοπτικές ε, μακροπρόθεσμες για να έχουμε και προοπτικές για οικονομική σταθερότητα. Παρατηρούμε με ενδιαφέρον το τι έκανε η Εστονία εδώ πέρα με μεγάλες δυσκολίες αλλά πάλεψε και δεύτερον σε ποιο βαθμό η διαρθρωτική μας πολιτική εδώ πέρα χρειάζεται να στηρίξει κάποιες ε, χώρες να εξειδικευτούν σε έναν τομέα όπως π.χ. η πληροφορική και εκεί πέρα να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ε, μια τόσο μεγάλη ικανότητα ώστε να προσελκύσουν παγκόσμιο ενδιαφέρον ε, των επενδυτών. Και εκεί πέρα βλέπω κάποια προβλήματα στην πολιτική συνοχής γιατί έχω την εντύπωση πως δίνουμε κάποια δισεκατομμύρια και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μόνιμη μείωση της ε, ανεργίας. Εάν δούμε κάποια κράτη-μέλη που η ανεργία είναι 35-40% εντελώς απαράδεκτο δηλαδή. Και γιατί, γιατί το βάρος ε, δίνεται κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν έχω τίποτα με τις μεγάλες επιχειρήσεις, σημαντικές κτλ. Καμία αντίρρηση, αλλά η λείπει μια μεσαία δομή και πολλές αυτόνομες ε, δομές σε ένα μέσο μέγεθος ε, επιχείρησης. Υπάρχουν ε, κάποιες επιχειρήσεις ενός ή δύο ατόμων, αλλά λοιπόν οι επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους. Οπότε γιατί τόση λίγη προσοχή σε αυτό ακριβώς το θέμα γιατί αυτά τα οποία θέλετε δεν γίνεται μόνο με τι οικονομίε, δεν είναι μόνο ο δρομο. Εγώ είμαι υπέρ τη οικονομία και τη αυστηρή οικονομία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, ληφθούν οικονομικά μέτρα για να έχει και μια προοπτική ο λαό ε, προ το μέλλον. Well, I that θα το θεωρήσω περισσότερο ως σχόλιο παρά ως ερώτηση. Ε, πιστεύω ότι οι περισσότερες πολιτικές ή δράσεις που ανέφερα, ίσως και δεν ανέφερα, αλλά εντάσσονται στις πρωτοβουλίες μας για την καινοτομία και την εσωτερική αγορά, εκεί ακριβώς αποσκοπούν. Γιατί ακριβώς αυτές οι επιχειρήσεις είναι αυτές που δημιουργούν απασχόληση, που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Θα έλεγα λοιπόν καινοτομία έρευνα, εκπαίδευση, δηλαδή διευκόλυνση συνεργασίας ε, και διαμεθοριακή κυκλοφορία μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, να δούμε το δυναμικό των αγορών. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που θα αν τις ανέφερα, είναι σημαντικές, είναι πολλές οι πρωτοβουλίες αυτές ε, και εκεί αποσκοπούν αυτό που θέλουμε να ενισχύσουμε στην ε, ενιαία αγορά και με την οδηγία για τις υπηρεσίες έχουν να κάνουν πολλά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρωτοβουλίες επίσης για τις δεξιότητες των εργαζομένων και νομίζω ότι όλα αυτά καλύπτουν ακριβώς αυτό το τομέα της οικονομίας πάνω απ' όλα. Κύριε θέλετε τώρα να μιλήσετε. Um, Έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω υπάρχει ο κίνδυνος ε, τα κράτη-μέλη εστιάζονται στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών και ταυτόχρονα είναι πολιτικά δύνατο να αυξηθεί ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα κινδυνεύουν και ο νομπελίστας ο κύριος Στίγκλιτς έχει προειδοποιήσει πως όλες αυτές οι περικοπές θα οδηγήσουν σε νέα ύφεση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν εάν είναι πολιτικά εφικτό ο προϋπολογισμός της Ένωσης να αυξηθεί για να χρηματοδοτήσει όλα αυτά τα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα για να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή ανάπτυξη. I think that I'm uh, not to... Δεν νομίζω ότι μου επιτρέπεται να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση. Αστιεύομαι. Νομίζω ότι ας το θέσω διαφορετικά. Θα έλεγα ότι υπάρχει κεφάλαιο όχι στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στις οικονομίες υπάρχει κεφάλαιο. Η Ευρώπη είναι πλούσια ήπειρο σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου. Το θέμα είναι πώς κινητοποιούμε το κεφάλαιο αυτό. Γιατί όταν μιλάμε για δημόσιο χρήμα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τους εθνικούς προπολογισμού. Εκτός μικροφώνου. Ναι, αν με ρωτήσετε προσωπικά, θα σας τα πω μετά. Γιατί αλλιώς ε, θα με καλέσουν στον τρίτο όρφο των Παρελεμών και θα με επιπλήξουν. Θα σας τα πω πολύ απλά, όχι σε οικονομικούς, με οικονομικούς όρους. Αν μιλάμε για δημόσιο χρήμα, τώρα εθνικό, κοινωνικό είναι χρήμα ε, δημόσιο, φόροι, φορολογία δηλαδή. Και φυσικά υπάρχει χώρος να συζητήσουμε κατά πόσον κάποιοι φόροι θα μπορούσαν να είναι πιο αποτελεσματικοί σε ενωσιακό ή σε εθνικό επίπεδο. Ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε περιθώρια βελτίωσης. Όπως είπατε από πολιτικής πλευράς δεν τίθεται καν, άρα ούτε καν το συζητάμε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά ποιο είναι ο περιορισμό, ότι πρόκειται για δημόσιο χρήμα. Επομένω, σε οποιαδήποτε περίπτωση, ακόμη και αν αλλάξει η σύνθεση και αυξηθεί ο κοινοτικό, ο ενωσιακό προπολογισμό, και πάλι θα πρέπει να δούμε πώ μπορεί να κινητοποιηθεί το ιδιωτικό κεφάλαιο. Και εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα στοιχείο αξιοπιστία. Όλοι δηλαδή φαίνεται σαν να περιμένουν να εξασφαλιστεί ότι δεν θα πάει τίποτα στραβά. Και αν σε πολιτικό επίπεδο η Ευρώπη είναι σε θέση, όπως το Μάρτιο περιμένουν, να έχουμε αυτό το συνολικό πακέτο που περιλαμβάνει τον χρηματοπιστοποιητικό και τον τραπεζικό τομέα, μόνιμος μηχανισμός, μεταρρυθμίσεις, ε, φραγκο, γαλλο, συγγνώμη, γερμανικές ιδέες κτλ αν εγκριθεί εγκαίρως το πακέτο για τη διακυβέρνηση. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο πακέτο αξιοπιστίας θα έλεγα και μπορούμε και εμείς να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο με αυτό για να κινητοποιηθεί και το ιδιωτικό κεφάλαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να θέσω ένα ερώτημα πριν ε, παραδώσω την, την Προεδρία. Πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο λοιπόν. Ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Στην Επιτροπή μας, στην ενδιάμεση έκθεσή μας, έχουμε κάνει τη διαπίστωση πως πρέπει να εμβαθυνθεί η ολοκλήρωση. Δηλαδή κοινό νόμισμα, κοινή νομισματική πολιτική χωρίς στενότερη οικονομική πολιτική, πολιτική ε, κοινωνική πολιτική και πολιτική προπολογισμού ε, αποδείχθηκε λάθος. Αλλά διαπιστώνουμε πως τα κράτη-μέλη παρά τα όσα λένε ε, στην πράξη καθυστερούν. Ξεκολουθούν να ακολουθούν την διακυβερνητική προσέγγιση δεν ακολουθούν την κοινοτική μέθοδο και δυσκολεύονται να αλλάξουν ε, αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό είναι το, το πρόβλημα. Όπως ακριβώς ε, και στον τομέα το χρηματοοικονομικό, το θέμα είναι η συμπεριφορά. Το βλέπουμε στα μεγάλα έργα ε, που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Όπως παραδείγματος χάρη ο Γαλιλαίος. Ο Γαλιλαίος είναι πέρα από το καλό και το κακό όπως είναι και το, ο τίτλος του βιβλίου, αν δούμε το τι ε, έχει ξοδευτεί από μεριάς χρημάτων. Γιατί, γιατί θέμε ένα ευρωπαϊκό έργο, θέμε πολλά εθνικά. Κάθε κράτος μέλος θέλει δικό του κέντρο ελέγχου. Έχουμε τρία κέντρα ελέγχου και μιλάμε για ανταγωνιστικότητα. Εάν είναι να κάνουμε έτσι τα έργα, ποτέ δεν θα έχουμε ανταγωνιστικότητα Οπωσδήποτε ε, δεν θα έχουμε διεθνή ανταγωνιστικότητα. Πρώτο αυτό. Οπότε το ερώτημά μου από τη δική σας τη Σκοπιά. Κοιτάξτε, εμείς ε, παλεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση, την κοινοτική μέθοδο δηλαδή, Κομισιό και Κοινοβούλιο. Αλλά στο Συμβούλιο υπάρχει ένας βασικός παίκτη που δεν θέλει ε, να παραδώσει τα, τα ενία. Ήμουν στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ ε, σε ένα πάνελ και εκεί πέρα είπα στους εκπροσώπους ε, του χρηματοοικονομικού τομέα πως δεν βλέπω καμία αλλαγή συμπεριφορά σας. Ε, συμβαίνουν τα συνήθη. Και είχα το, το αφελές όνειρο, την αφελή ελπίδα πως κάποια αλλαγή συμπεριφοράς θα, θα υπήρχε. Και υπήρξε κάποια σιωπή από κάτω και είπα πως εγώ στη δική σας θέση τα μπόνους τα οποία πληρώνετε όπως τα υπολογίσατε αλλά τα μπόνους ενός έτους και πιθανώς δύο ετών να μην τα πληρώσετε αλλά να τα πάρετε και να χρηματοδοτήσετε ένα έργο παραδείγματος χάρη για την ανεργία των νέων. Μιλάμε για δισεκατομμύρια, γιατί είναι διψήφιοι αριθμοί δισεκατομμυρίων. Εάν είχε πει όλος αυτός ο κλάδος φέτος το 2009 δεν θα δώσουμε μπόνους, θα τα υπολογίσουμε και τα λεφτά θα πάνε σε ένα ταμείο το οποίο θα λέγεται ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Απασχόληση των Νέων. Ξαφνικά θα είχαμε 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Σιωπή παγωμένη, γιατί οι κυρίες και κυρίοι, υπήρχαν και κυρίες, δεν σκέφτηκαν για ένα δευτερόλεπτο κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι το χειρότερο. Δυστυχώ αυτό συμβαίνει και αυτό συμβαίνει και αυτό ισχύει και για τα κράτη-μέλη. Ε, ο Γαλλίος είναι σχεδόν παρελθόν, αλλά σας εγγυώμαι, το επόμενο έργο θα γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα γίνει με ευρωπαϊκό πνεύμα, αλλά ποιο κομμάτι του έργου μπορώ να πάρω εγώ και α γίνει δύο και τρει φορές. Και ε, πλέον, ναι, δεν, είναι, δεν θα είμαστε διεθνώ ανταγωνιστικοί. Νομίζω αυτή είναι ερώτηση αρμοδιότητας ψυχιάτρου. Νομίζω συμφωνούμε. Ήταν περισσότερο σχόλιο παρά, παρά ερώτηση. Απλά ήθελα, ήθελα να το πω. Ναι, ναι, το, το βλέπω σε, Είναι θετικό αυτό. Νομίζω συμφωνούμε με τα περισσότερα από αυτά. Ε, κάποιες φορές ε, προξενεί έκπληξη το ότι στην ε, κατάσταση αυτή της κρίσης βλέπουμε αύξηση της διακυβερνητικής προσέγγισης. Αυτό το οποίο θα έλεγα είναι πως πρέπει πραγματικά να κάνουμε μια προσπάθεια από πλευράς θεσμικών οργάνων να έρθουμε σε επαφή με τον έξω κόσμο όπως είπα, αν στείλουμε όλα αυτά τα έγγραφα, αν δούμε τις πολλές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν από πλευράς Κομισιόν το Μάιο του 2010, εάν τα δώσουμε αυτά σε οποιονδήποτε, ακόμα και άτομα ε, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είπε κάποιος, ε, χανόμαστε, δεν ξέρουμε τι, τι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε έχουμε μία ευθύνη, νομίζω, να πετύχουμε την ουσία και να εστιάσουμε στις προτεραιότητες και μετά τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα σε καιρούς κρίσης. Αλλά αυτή η, η, αίσθηση της συλλογική ευθύνη έπρεπε να είναι πιο, πιο έντονη. Σαν τις Πρεσέδο. Ευχαριστώ πολύ. Όταν μίλαγε ο πρόεδρος θυμήθηκα κάποιους που λένε ότι είναι πιο εύκολο να δεχθεί κανεί νέε ιδέες παρά να εγκαταλείψει παλές πρακτικέ. Και νομίζω ότι αυτό το βλέπουμε και το επιβεβαιώνουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω με τη στρατηγική 2020, όπως και με όλες τις ε, πρωτοβουλίες οι οποίες προτείνονται τελικά, η εντύπωση που αποκομίζει κανείς είναι ότι είναι ένα σύνολο εγγράφων που θα θεσπίσουν κάποιες πρακτικές, αλλά τελικά ε, δεν έχουμε αποτελέσματα αλλά προβλήματα και είναι ουσιαστικά ένα ζήτημα αποτελεσματικότητας πάνω απ' όλα. Σήμερα τίθεται η ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σε καλή κατάσταση τα δημόσια οικονομικά για να υπάρξει όμως δημοσιονομική εξυγίανση και ταυτόχρονα αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ερωτώ, από πού θα έρθουν οι επενδύσεις, ποιες είναι οι νέες πηγές χρηματοδότησης από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια θα μπορούσε να πει κανεί τελικά ότι τα δημοσιονομικά, τα φορολογικά από έναν ξεκινούν, από τον πολίτη. Ο φορολογούμενος είναι αυτό που πληρώνει, που πληρώνει του φόρου, Αλλά ξέρουμε ότι ε, υπάρχουν μεν διαφορετικές ε, αναχώρα φορολογικές πηγές, ε, αλλά δημιουργούνται προβλήματα από αυτές και θα πρέπει, είναι ένας πολύ λεπτό τομέας αυτός του κεφαλαίου, δημοσιομικός, ο χρηματοπιστωτικός, επιχειρήσεις, αλλά πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προοδεύσει, να σημειώσει κάποια πρόοδο στον τομέα αυτό. Κάτι άλλο που συζητείται διαμακρών σήμερα είναι η σταθερότητα, οι διαφορές, το σύμφωνο ανταγωνιστικότητας. Όταν μιλάμε για τους μηχανισμούς σταθερότητας, αυτοί που πρέπει να δώσουν εγγύησεις, προσπαθούν πάντοτε να μην έχουν μεγαλύτερα πλεονεκτήματα ε, από κοινωνική πλευρά και να κάνουν λιγότερη δημοσιονομική προσπάθεια. Εμεί θέλουμε όμω να υπερκεραστούν οι διαφορέ αυτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει και στο κοινωνικό και στο φορολογικό και στο δημοσιονομικό τομέα. Και δεν μπορούμε μόνο να έχουμε ως προοπτική τη μείωση του εργασιακού κόστους, θα πρέπει να έχουμε και ένα ε, κατώτατο όριο, δηλαδή να θεσπίσουμε κάποια κατώτατα, κάποια ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα. Και έχω την εντύπωση ότι ουσιαστικά ε, κάπως ε, σφίγγουμε τις βίδες ε, και κάνουμε κάποια έτσι μικρή διόρθωση, αλλά δεν κάνουμε τίποτε περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τώρα τα διάφορα θέματα που ετέθησαν, σε ό,τι αφορά την ψηφιακή ατζέντα θα ήθελα εγώ να, να πω κάτι. Σημαντικό, σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι στη ΣΥΠΑ λαμβάνονται αυτή τη στιγμή όλες οι πρωτοβουλίες. Ξεκινήσαμε καλά στην Ευρώπη με τις τηλεπικοινωνίες, αλλά κάπως χάσαμε το βηματισμό μας, θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρουμε προς τα πού να πάμε τώρα, πώς να συνεχίσουμε. Το ζήτημα τώρα της ανάπτυξης, εσωτερική αγορά, αλλά οι αναλυτές μιλούν για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και λένε ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση τα επόμενα δέκα χρόνια, θα τριπλασιαστεί συγκεκριμένα στι αναδυόμενε οικονομίε. Αυτό δεν θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και μια πολύ στέρεη και συνεπή στρατηγική και για το εξωτερική στρατηγική. Και επίσης, ποιος είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει η Ευρώπη στο παγκόσμιο προσκήνιο. Όταν πρέπει να λαμβάνουμε σε πραγματικό χρόνο αποφάσεις, είμαστε κατακαιρματισμένοι και αυτό πραγματικά ε, είναι κρίμα ε, στην διεθνή σκηνή εικόνα που δίνει η Ευρώπη. Αυτά, θα ήθελα ένα σχόλιο για όλα αυτά που είπα. Ευχαριστώ. Για πολλά από αυτά τα θέματα. Ουσιαστικά καλύψατε ένα ευρύ φάσμα, μάλλον επί παντός επιστητού μιλήσατε θα έλεγα. Για τη σχέση μεταξύ την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την εξυγίαση των δημοσιονομικών και από πού πρέπει να έρθει το κεφάλαιο, το γεγονός ότι αναδιαρθρώνεται ή θα έπρεπε να αναδιαρθρώνεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο σε θέση να χρηματοδοτήσει την οικονομία. Αντίθετα, αυτό θα πρέπει να βοηθήσει τις τράπεζες να είναι πιο ικανές να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία. Το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερα. Αυτή η αηδία που έχουμε, έχουν ορισμένοι για τον κίνδυνο, αυτή η έλλειψη αξιοπιστίας, αν αυτό ξεπεραστεί, θα επανέλθει δρυμύτερο ο χρηματοπιστωτικό τομέα. Γιατί δεν το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Υπάρχει πολλή ρευστότητα. Απλώ κάθονται τα λεφτά κάθονται κάποιοι πάνω στα λεφτά. Δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ τη αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη ικανότητά του να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία. Αντίθετα, νομίζω ότι γίνεται και είναι θετικό στοιχείο να, μπει, να φτάσει σε θέση που να μπορεί να το κάνει, να θέλει μάλλον να το κάνει. Τώρα για την ενιαία αγορά. Πρέπει να την ε, συνδυάσουμε και την, να δούμε και την ε, εξωτερική διάσταση, την εξωτερική αγορά. Θα πρέπει οι εταιρείε μας να είναι σε θέση να πάνε και προς το εξωτερικό και μέσω της ε, εκμετάλλευσης των θετικών στοιχείων της εσωτερικής αγοράς οι εταιρείε ενισχύονται και είναι έτοιμες για να βγουν προς τα έξω. Φυσικά, η, η ζήτηση ευρωπαϊκών προϊόντων προφανώς θα προέλθει κυρίως από τις αναδυόμενες οικονομίες. Παρ' όλα αυτά το εμπόριο το ενδοκινοτικό δεν είναι μικρό, δεν είναι αμεληταίο, αλλά το επιπλέον το έξτρα θα είναι μεγαλύτερο απ' έξω πια. Αλλά μην ξεχνάμε και το, εσωτερικό, και το εσωτερικό εμπόριο, το ενδοκινοτικό. Παραδείγματο χάρη για τη Γερμανία είναι 20%. Και μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία είναι μεγάλη εξαγωγική χώρα. Ε, είναι ακόμα σημαντικό στοιχείο η ενιαία αγορά. Το να δώσουμε έμφαση τώρα στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και στο ψηφιακό τομέα, ναι, συμφωνώ. Υπάρχουν διάφορε σχετικέ πρωτοβουλίε και νομίζω ότι στα πλαίσια τη Ευρώπη του 2020 υπάρχει ένα κεφάλαιο με μια δέσμη πολιτικών για το θέμα αυτό. Για την κατανομή και την εξέλιξη των μισθών, Οι μισθοί θα πρέπει να εξελίσσονται ανάλογα με την παραγωγικότητα. Φυσικά πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες για τις ευπαθείς ομάδες και υπάρχει αυτό και στις πολιτικές μας. Εδώ αυτό συνδέεται με τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα, με την ελάχιστη κοινωνική κάλυψη Συγκλήσεις και αποκλήσεις. Για κάποιες χώρες υπήρξε μια περίοδος υπερβολικής σύγκλησης, αλλά δεν είχε στερεά βάση. Γι' αυτό υπάρχει εκ νέου μια απόκληση. Ε, αυτό δεν είναι γενικευμένη τάση, αφορά μερικές χώρες. Είδαμε μια πολύ γρήγορη σύγκληση για κάποιες χώρες, ιδίως εκείνες που επωφελήθηκαν από τη φούσκα των ακινήτων και είχαμε τρομακτική αύξηση των μισθών και τώρα βέβαια πέφτουν στον αδύρ οι μισθοί. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος να τη ζήσει κανείς, αλλά είμαστε σε φάση εξισορρόπησης. Μιλάμε για μισθούς, δηλαδή οι οποίοι δεν ήταν βιώσιμοι, δεν μπορούσαν να συνεχιστούν σε αυτό το επίπεδο. Θα διανύσουμε μια περίοδο απόκλησης λοιπόν, αλλά οι χώρες που είναι ουραγοί θα κινηθούν πιο γρήγορα. Θα υπάρξει δηλαδή εκ νέου μια τάση σύγκλησης. Ευχαριστώ. Βλέπω πως δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος τον λόγο. Οπότε θα ήθελα κυρία Φλαούρας να σας ευχαριστήσω για το ότι ήρθατε εδώ πέρα για να μιλήσετε εξ ονόματος της Κομισιόν και να μιλήσετε τόσο ανοιχτά και με ειλικρίνεια για όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ.